Καλημέρα σε όλους και όλες αγαπητοί συνάδελφοι. Να βρούμε όλοι μας από μια θεσούλα και να προετοιμαστούμε για αυτό το πρωινό που θα είναι γεμάτο ψηφοφορίες και να το κάνουμε ήρεμα γιατί θα έχει πολλές ψηφοφορίες γι' αυτό μήπως θα μπορούσαμε να σιωπήσουμε και να σεβαστούμε το χώρο. Ε. Audi. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η ψηφοφορία σήμερα και θέλω να γνωρίζω κατά πόσον τηρήθηκαν οι κανόνες πολυγλωσσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν μέρη, εν μέρη. Έχουμε τις γλώσσες όλες αλλά όχι Μάλτας και Εσθονίας. Αυτές οι δύο γλώσσες μας λείπουν. Θα ήθελα να υποβάλω μια ένσταση για την υποβάθμιση της πολυγλωσσίας στο Κοινοβούλιο, ιδίως για σημαντικά κείμενα τα οποία θα ψηφίσουμε. Διότι ουσιαστικά πρόκειται για άσκηση της πολιτικής εντολής που μας έχει ανατεθεί και θέλουμε να υπάρχει και πρόσβαση των πολιτών στο έργο μας. Άρα σας παρακαλώ να γραφεί η ένστασή μου στα πρακτικά. Η πρόεδρο είναι τα γραπτά κείμενα δεν υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες. Ναι, εντάξει, η γραμματεία θα τα συμπεριλάβει στα γραπτικά. Λοιπόν, η μερίσια διάταξη τώρα την έχετε. Ξεκινάμε αμέσως τις ψηφοφορίες μας. Άρθρο 70 αναθεωρημένο του κανονισμού. Αν δεν έχετε κάποια παρατήρηση να κάνετε, τότε χωρίς αλλαγές ε, υιοθετείτε η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, οι Μαλτέζοι και οι Εστονοί δεν θα ακούνε στη γλώσσα τους, όλοι οι υπόλοιποι ναι. Ελπίζουμε να μην είναι, να είναι γοργή όλη η διαδικασία, ίσως και πέντε λεπτά μια παύση να κάνουμε μετά από το σύνολο των τροπολογιών Έλλερ. Εντάξει, και μετά πάντως μετά από κάθε θέμα που θα εξετάζουμε θα έχουμε μια σύντομη διακοπή για να ξεκουραστούμε λίγο. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό να κάνουμε ένα έλεγχο, να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματά μας. Σας παρακαλώ για να δούμε. Ψηφίζουμε για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματά μας. Tutti avete votato sì. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω είναι. Ναι, τώρα, τώρα, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τέλος της ε, δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Πάμε παρακάτω τώρα. Ψηφίζουμε ακριβώς το κείμενο για την έκθεση Μαντουρέλ. Συμβαστική λύση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το γυναικών 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 και 456 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 457 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 458 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 459 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Α, όχι. 48-48 όχι λοιπόν. Καταπίπτει. Συμβαστή 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 534 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική λύση 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 508 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική λύση 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 523 το δεύτερο μέρος. 523 παραλαμβάνω, δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές. Κανονικά απορρίπτεται να ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά. 523 δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 527 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 526 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 συμβαστική λύση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 529 και 534 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 405 και 431 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 574 και 15 υπέρ κατά αποχές. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 574 και 15 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά εκεί στο βάθος δεν 574 και 15 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ Πέρες ψηφοφορίες απορρίπτεται. 27-27. Ισοπαλία και απόρριψη. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω. 548 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16. Α, μισό λεπτό, μισό, ε, μισό λεπτό. Τόγια. Κυρία Τόγια. 16. Υπέρ. Κάπως είχαμε μπερδευτεί. Λοιπόν, άφετ 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική λύση 16. Στην άφετ 16. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Votazione chiusa. Πέρας τη ψηφοφορία. 16 και πριν από τη συμβαστική 16 ποιος έχει το λόγο. Κύριε Τόγια. Πρόεδρε, η τροπολογία μου 581 να αποσυρθεί, την αποσύρω, γιατί δεν καλύπτει συμβαστική λύση, άρα λοιπόν ε, την αποσύρω. Ευχαριστούμε κυρία Τόγια. Ψηφίζουμε τώρα την συμβαστική 16 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 585 υπέρ, ε, συγγνώμη, 565 ε, υπέρ κατά. Δικαστήριο. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Δεν ακούμε. μπορούμε να παρακολουθούμε τις τροπολογίες. Ε, σας παρακαλούμε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί καθυστερούμε λόγω της μετάφρασης. Δηλαδή, μετά τις συμβαστικές, δώστε μας λίγο παραπάνω χρόνο, μην τα λέτε τόσο γρήγορα. Perfetto. Ωραία. 565 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 566 και 43 μαζί υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 570 και 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 572 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 573 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 575 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ, 575. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 586 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 577 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 588 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, 9, 7 και 10 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας από το ΕΛΚ ε, είναι παραπάνω. Συνεχίζει να είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. 26-26 και απορρίπτεται. 457. Υπέρ. Κατά. Τετρακόσια, 474 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 473 και 32 3 ε, μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 636 και με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 636 ηλεκτρονικά παρακαλώ με την προφορική τροπολογία. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. 30-23 εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 και 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 685 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20... Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για την 685 ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Από το ΕΛΚ είναι ένας παραπάνω και πάλι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. 26-26 πάλι απορρίπτεται. «24 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται». Η 687 υπέρ, κατά, αποχές. Κανονικά εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και σε αυτό παρακαλώ. είναι μισές μισές οι προτιμήσεις, γι' αυτό είναι δύσκολο να το βλέπουμε καθαρά από την αρχή. Πέρες φιοφορίες. Α, εδώ 31-23 εγκρίνεται. 62, 692 και 4 και 3 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 688, 689, 690, 16, 54, 691. Αυτές όλες μαζί. Αλλά σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 Η γραμματεία μου λέει... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για να δούμε. Ποια μένει απ' έξω. Συγγνώμη, λάθος, λάθος. Κάναμε λάθος. 691 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μαζί τώρα οι 693 και 695 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας 28-26 εγκρίνεται. Η 694 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, έχουμε τα κείμενά μας λίγο που μας μπερδεύουν. Συνεχίζουμε. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 697 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 698 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 18. Όχι. Όχι. Η 699 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 700 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 702 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 705 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 706 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 711 και οι 56 μαζί αυτές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 713, 714, 37, 55 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 712 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 715 υπέρ. 715. Τσουκάλας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. MV57 υπέρ. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 726 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ 41. Ναι, να ελέγξουμε για τη 41 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Απορρίπτεται. 39 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 727 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 31-22 εγκρίνεται. 7-28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 740 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 και 741 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 και 742 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 και 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 752 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 754 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 775 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 758 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 759 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 778 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 886 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 886. Πέρασε. πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 909 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 928 με προφορική τροπολογία υπέρ 928 λοιπόν προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 989 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 997 τροπολογία. 997 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μήπως να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 997. Πέρα της ψηφοφοριας 32.21 32-21 εγκρίνεται. 44 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1042 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1061 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέξουμε 1061 και ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Για να δούμε. Α, εντάξει τώρα, εγκρίνεται. 33-22 το αποτέλεσμα ήταν. Συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1212 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 33-22. Εγκρίνεται. 1220 υπέρ. Κατά. 1220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1224 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1271 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ναι, είναι σαφές το αποτέλεσμα. 26-28 και μόλις απορρίφθηκε. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43, συγγνώμη, 53 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. περας ψηφοφοριες ψηφοφορίας. 27-28 απορρίπτεται για μία ψήφο. «1295 υπέρ, κατά, αποχές». Βλέπω ότι είμαστε πάντα μισή-μισή, γι' αυτό σας παρακαλώ και πάλι ηλεκτρονική ψηφοφορία να ελέγξουμε. 1295. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. επιμένει, επιμένει ο ένας ο παραπάνω από το ΕΛΚ. Κανείς, <laughs> κανείς δεν αποχωρεί. Τώρα εντάξει. 30-24 και εγκρίνεται. 1278 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1322 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέξουμε, να ελέξουμε. Από τη στιγμή που το ζητάτε θα σας ικανοποιήσουμε. Πάλι ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Επιμένει ο παραπάνω από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί. Επιμένει. Πέρας ψηφοφορίας. 28-27 για μία ψήφο περνάει. Εγκρίνεται. 1337 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1337 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίζουμε. 25-29 και απορρίπτεται. 54 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 συμβαστικοί υπέρ. «55 συμβαστικοί. Μπορείτε να βρείτε την 55 και να ανταποκριθείτε. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1485, υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι 1485 πάλι ο παραπάνω από το ΕΛΚ επιμένει αποσύρθηκε εντάξει 27-23 και εγκρίνεται 56 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1686 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Κανονικά εγκρίνεται αλλά να σιγουρευτούμε. Πέρας ψηφοφορίας. 27-28 απορρίπτεται για μία ψήφο. Απορρίπτεται. 1740 υπέρ κατά αποχές κανονικά απορρίπτεται να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά εσείς λέτε περνάει εγώ λέω απορρίπτεται να δούμε ποιος έχει δίκιο Πέρας ψηφοφορίας. 28-27 εγκρίνεται για μία ψήφο. 1742 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Επιτρόπο. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Α, δύο από το ΕΛΚ παραπάνω αυτή τη φορά. φοβοριες ψηφοφορίας. 25-28 και απορρίπτεται. 60 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά στην προηγούμενη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Εντάξει.

Η 222 απο... αποσύρθηκε. Λοιπόν, τροπολογία 228 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 64 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 65 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ένα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 241 σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές να το ελέξουμε ηλεκτρονικά το. Πρώτο μέρος λοιπόν του, της 241. Πέρας ψηφοφορίας. 27-27. Άρα λοιπόν απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Άρα σε αυτό Αφετ 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 242 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρανς 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 Γεωργίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 262-263 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 264 και 9 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προπολογισμού 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 και 295 με προφορική επιστροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέξουμε για τη 13. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Votazione. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 26-30 απορρίπτεται η 13. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 8, 17 και 286 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, 19. Ψηφίσαμε για αυτήν. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13 να ελέγξουμε για τη 12, εντάξει. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη 12 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίες Απορρίπτεται. 23-33. 13 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανονικά εγκρίνεται να το ελέγξουμε όμως. Οριακά είναι. Για να δούμε. Πέρας ψηφοφορίας. 23-32 απορρίπτεται. 14. εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 Εντάξει, η προηγούμενη ε, κανονικά μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Να το ελέξουμε ομω Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ναι, ναι, εγώ έκανα λάθος λέει η πρόεδρος. 3.16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να δούμε τι εννοείται. Θέλετε να ελέγξουμε, όχι, όχι. 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 6 αφέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η κατά 21 ψηφίζουμε την προηγούμενη ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 33 21 21 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Ναι, ελέγχουμε για το δεύτερο μέρος λοιπόν. ψηφοφορίες ψηφοφορίας. 24-32 και απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 354 355 359 14 και 22 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 82 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 372 υπέρ, κατά αποχές να ελέξουμε ηλεκτρονικά. 372 λοιπόν ψηφίζουμε. Πέρασε. Και πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. 34-21 και εγκρίνεται. 20 και 19 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 και 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Κανονικά απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε. Έτσι. «28-28 και απορρίπτεται». 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. 55 και μία αποχή. Τέσσερις ψηφοφορίες για το ψήφισμα. Προπολισμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προπολισμός 3 περ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα και ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Υπέροχα. 55 με μία αποχή.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 Abbiamo deciso che la pausa la facciamo dopo Eller, no? Με, μετά από το επόμενο θα κάνουμε το διάλειμμά μας, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Καρβάλιο. Prego. Cominciamo con un voto in blocco NV5 ed NV6. A favore? Contrari? Astenuti? Respinto. Altro voto in blocco. Λοιπόν, 185, 195, 196, 458, 460, 978, 161 στο σύνολό τους υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 3 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, οι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, οι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, οι 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 3α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 232 υπέρ κατά αποχές Προλαβαίνω να ακούσω τη μετάφραση. Σας παρακαλώ, πιο σιγά. Έχουμε κάνει δουλειά μηνών, μην τη χαλάσουμε έτσι. Η κυρία λοιπόν διαμαρτύρεται ότι δεν προλαβαίνει. Δύο τριανταδύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Compromesso 3B. A favore. contrari. Η επόμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Emendamento 19. A favore. Η επόμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 235 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.38, 2.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.42, Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επόμενη η 2.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.42 υπέρ 2.52 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2.52 2.52 ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ε, chiuso. 28 29. 28-29 απορρίπτεται για μία ψηφοδιαφορά. 2-52. 2-46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2-53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 2.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το σύνολο τώρα 2.56, 2.58, 2.57, 2.60, 2.59 και 2.62. Μαζί όλες αυτές υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 261 υπέρ. Πώς είπατε. La girava Τι γίνεται διάφορες φωνές και διαμαρτυρίες στην αίθουσα. Άδικο είχα, άδικο είχα. Είχαμε ψηφίσει ήδη στο σύνολο τη 261. Άρα λοιπόν τη 263 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 264 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 5 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 326 το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η, η 600 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Να ελέγξουμε για την 600 ηλεκτρονικά. Pepe di troppo. Pepe Πέρας. 38-17 και εγκρίνεται. 12 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 919 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 920 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 601 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 608 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέξουμε 608 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Votazione chiusa. Πέρας. 27-29 και απορρίπτεται. 6-19 υπέρ. Μήπως την ψηφίσαμε την 6-19. 6-19 ψηφίζουμε. Κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 6-19 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 27-29 και απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν η 6-19. 22 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «701 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». 23 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 688 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέραση ψηφοφορίας και ψήφισαν όλοι, πέρας. 28-25 εγκρίνεται. 24 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 979 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 980 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 981 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 982 υπέρ κατά αποχές Κανονικά εγκρίνεται να το ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά. Πέρασε. 29-26 εγκρίνεται. 9-83 83 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε και εκεί. Πέρας. 24-31 απορρίπτεται. 27α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τη συμβαστική. Έμβη 113, 116, 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμβη 114, 117, 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκριένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, MV1 η προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΦΑΜ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η ΦΑΜ ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τέσσερα τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΦΑΜ δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι είχε καταπέσει αυτή, δεν ίσχυε πια. Α, λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1α συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 32-23 και εγκρίνεται. Καλτένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγκριτρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλτ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα, ένα μπι συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές 183 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για 183 όχι όχι, όχι. Ε, με ένα τασχυρός λοιπόν τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας 55-0 εγκρίνεται ομόφωνα και ψηφίζουμε για την ε, νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 53 και ένας κατά. Συγχαρτήρια. Συνάδελφος Καρβάλιο, συγχαρτήρια. Αυτά. Και τώρα, Χέλερα. Και μετά, μετά, μετά θα διακόψουμε λίγα λεπτά για να ξεκουραστούμε, να απαυθούμε. Allora. Και αν είμαστε έτοιμοι. Έλερ. Έλερ, έλερ. Allora. Λοιπόν, 177 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, για να δούμε. Βλέπουμε ο κόσμος εδώ, αγκαλιάζεται στους διαδρόμους, φιλιέται. Να τελειώσουν λοιπόν και ψηφίζουμε. 177 ψηφίζουμε μετά από τους εναγκαλισμούς. Ψηφίζουμε. Πέρας. 23-28 απορρίπτεται. 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188-191 μαζί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 και 2.30 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέξουμε ηλεκτρονικά. Ε, Χιούζα. Πέρας ψηφοφορίας. 24-31. Απορρίπτεται. 2.45 και 14 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.45 και 14 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας απορρίπτεται. Δύο και 15 μαζί. 2.47 και 15 υπέρ, κατά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, όχι, καταπίπτουν αυτές, άρα λοιπόν δεν ψηφίζουμε. Άφετ 2. Καταπίπτουν οι υπόλοιπες. Αφετ 2. Αφετ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.50. Μαζί και 31. Όχι 31. Υπέρ. Τι γίνεται με αυτές. Καταπίπτουν μήπως. Ναι, ναι. Εδώ από δεξιά μου λένε ότι είναι ψηφίσμε. 31 λοιπόν, 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.46 και 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. αφετρία υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την αφετρία Πέρας. 28-26 εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 269 και ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 29-24 εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.71 υπέρ κατά αποχές κανονικά εγκρίνεται να το ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά έτσι για να σιγουρευτούμε Κιούζα Περάς εγκρίνεται 27-25 εγκρίνεται 2.72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.98 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά και σε αυτό. Πέρας. 27-28 μόλις μόλις απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.78 υπέρ κατά αποχές που απορρίπτεται. 278 ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Και Α, ένας παραπάνω από το ΕΛΚ πάλι. Λοιπόν, πέρας. 26-26. Καταλαβαίνετε λοιπόν, απορρίπτεται. αλλάζει το αποτέλεσμα. 27-26 μόλις μόλις εγκρίνεται. 24 συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλερ. 278. Um, I understand it. Για την 278 κατάλαβα πως ήταν 26 με 26 η ψηφοφορία. Ναι, ακούστε, ακούστε, να ξαναψηφίσουμε αν θέλετε, αλλά εδώ ο συνάδελφος μου είχε πει ότι δεν είχε μπορέσει να ψηφίσει, προσθέσαμε την ψήφο του και πήγαμε 27-26 για να ξαναψηφίσουμε. Λειτουργεί το μηχάνημά σου. Ναι. Λοιπόν, 2.78 ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 2.78 ξαναψηφίζουμε. Πέρας. 28-26 τώρα. Κερδίσαμε και μία ψήφο. Λοιπόν, εγκρίνεται. 24 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 293 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 297 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ παρακαλώ λίγη ησυχία για να μην μπερδεύομαι κι εγώ που είμαστε, σε ποια είμαστε 2.97 πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.33 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Σκίνερ. 3.33. Τελειώσαμε. 25-30 απορρίπτεται. 3-39. Α, μισό λεπτό. 26 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3-39. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3-45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού είμαστε? 3.45 ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. ...3.45 πέρας... ...30.25 εγκρίνεται... ...27 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται... 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 375 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 381 και 382 μαζί υπέρ κατά τι, τι γίνεται εδώ ελέγχουμε 381-382 ελέγχουμε ηλεκτρονικά 381-382 Πέρας ψηφοφορίας 35-19 εγκρίνεται. Αφετ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 390 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 32 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 412 υπέρ, 412, 412, πρώτη 412 υπέρ. Το βρήκατε στα κείμενά σας. Εντάξει. 412 πρώτη ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 417 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 471 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 474 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 474 πέρας ψηφοφορίες 21-34 απορρίπτεται. 33 συμβαστική υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 478 υπέρ κατά. Αποχές κανονικά απορρίπτεται. απορρίπτεται. 4-84 και με την ΑΦΕΤ 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 συμβαστική και 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 493 υπέρ κατά αποχές να ελέξουμε ηλεκτρονικά. Να ψηφίσω κι εγώ ή όχι. Εναντίον σου ψηφίζεις. Ε, θα μας εξηγήσει μετά τι συμβαίνει. Συγγνώμη, λάθος. Λάθος. Ένα υπέρ, δύο υπέρ τώρα, ναι. 493 απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5.24, 5.25, 5.26 μαζί αυτές υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις τρεις. Εντάξει. 524, 525, 526 ψηφίζουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 16.38 απορρίπτονται. 5.27. 5.27 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 528 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 547, 548, 549 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 38 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. 39 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 558 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 559 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 601 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 613 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 συμβαστική υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 συμβαστική υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, έκανα λάθος, λέει πρόεδρος, το 42, φαίνονταν καθαρά εντάξει, αλλά μου ξέφυγε, μου ξέφυγε, εγκρίνεται. Λοιπόν, η 42 είπαμε εγκρίνεται. 43 συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 663 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 674 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές κανονικά εγκρίνεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 92 Έλερ. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. εξακολουθεί να επιμένει ο παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας. 40-14 εγκρίνεται. 6-96 και 39 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 705 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 τώρα. 706-707 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 708 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 756 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 749 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 763 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 764 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Να ξεκουραστούμε κιόλα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 764. Πέρασε. 3122 και εγκρίνεται. 53 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ποια να ελέγξουμε. Τη συμβαστική, 53 τη συμβαστική ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 53 συμβαστική ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Η μία. Λοιπόν, πέρασε. 33-22 εγκρίνεται. Μαζί τώρα. 742 και ντεβε 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 743 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 766 υπέρ κατά να ελέγξουμε ελέγχουμε Αυτή τη φορά δύο παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει, ρυθμίστηκε. Πέρας. 33-21 και εγκρίνεται. Ένα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 έλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 έλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές κανονικά απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. 29-24 και εγκρίνεται. 5 συμβαστικοί και 6 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστικοί 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές κανονικά απορρίπτεται να ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά παρακαλώ. 143 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ, η μία. Πέρας απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. 15-40. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 Λάμπερτς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας λοιπόν. 16.38 απορρίπτεται. 158 και ντεβε 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή μήπω όχι. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 172 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Πέρας. 27-28 απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. DV6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. βέβαια 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. 51 υπέρ, αποχές 3 για τον ε, εισηγητή συγχαρτήρια. Ψηφίζουμε το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ, πέρας της ψηφοφορίας. 52, μία αποχή. 52-1. Παρακαλώ, 10 λεπτά, 10 λεπτά διάλειμμα. Διακόπτουμε για 10 λεπτά, έτσι. Και μετά ξεκινάμε και πάλι. Σα ευχαριστώ για τη συνεργασία σα. Για 10 λεπτά διάλειμμα, λοιπόν. Bene, prendiamo posto. Proseguiamo il nostro. Ξεκινάμε και πάλι. Allora, collega Odi ha chiesto la parola, prego. Odi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με την παρατήρηση που έκανα πριν για την πολυγλωσσία και για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν μίλησα για τη διερμηνία και την μετάφραση των ε, εγγράφων, αλλά μάλλον για την μετάφραση των εγγράφων τα οποία είχαμε υπόψη μας για τις ψηφοφορίες. Αναφέρομαι στα γραπτά κείμενα. Εντάξει, εντάξει, το είπαμε προηγουμένως, ε, το βάζουμε λοιπόν στα πρακτικά ότι εννοούσε ο κύριος Φοντή την γραπτή μετάφραση και όχι την ε, προφορική διερμηνία. Φιλίπ Λαμπέρ. Έκθεση Λαμπέρ. Κάτι μικρό για τα πρακτικά και συγχαίρω τους τρεις εισηγητές. Υπήρχαν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες όπου βάλατε το όνομα του ECR αλλά δεν τις είχαμε στηρίξει. Ε, απλά το διευκρινίσα για τα πρακτικά. Μάλιστα, θα το, θα το ελέγξουμε. Ωραία, πολύ καλά. Έτοιμοι όλοι. Ψηφίζουμε και πάλι. Έτοιμοι, έτοιμοι. Λοιπόν. 16 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κάλτε 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 και καλτ ε, μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό να ελέγξουμε. 23, 23 ελέγχουμε και, και 10. Ε, ναι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε λοιπόν. Και αν ψήφισαν όλοι. Λείπουν μερικοί όμως. Πέρας. 22-25 απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 19 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 119. Ψηφίσαμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές κανονικά απορρίπτεται να το δούμε όμως ηλεκτρονικά. Δεν είχατε ψηφίσει. Για να δούμε λοιπόν. αν ψηφίσαμε. 21-25 απορρίπτεται. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36, 56, 57, 58. Όλες μαζί ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 46 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μαζί 152, 153 με προφορική υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Κάλτ 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή η συμβαστική. 25 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ελέγχουμε για τη 18 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 25-24 εγκρίνεται για μία ψήφο. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές. Πώς είπατε? Ψηφίζουμε και πάλι. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλτένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τρία συμβαστική υπέρ, κα, συμβαστική τρία είπαμε, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά συμβιβαστική. Πέρας ψηφοφορίας. 25-24 εγκρίνεται. 4 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πέντε συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζούρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές Κανονικά εγκρίνεται να το ελέξουμε όμως. 86 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 22-23 απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλτ 5 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε καλτ 5 πέρας 27-22 εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέξουμε, να ελέξουμε. 97 ελέγχουμε για την 97. Πέρας. 23-23 απορρίπτεται μοιρασμένη η ψηφοφορία. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάζετ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές Κανονικά εγκρίνεται να ελέξουμε ηλεκτρονικά. 169. Ελάτε στα γρήγορα. Πέρας. 30-21 εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174. Μισό λεπτό, μισό λεπτό όχι, τζούρι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174. Λοιπόν, 175 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 175. Πέρας. 21-30 απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζούρι 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 181 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 25-26 απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αυτή. Αμφιβάλλεις Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 184. 184 περας πέρας. 24-26 απορρίπτεται. Τζούρι 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 22-29 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. 46 υπέρ, 4 οι αποχές εγκρίνεται. Λάμπερτ, ε, συγχαρτήρια, ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας. 44 υπέρ. Συγχαρτήρια. Τώρα έκθεση Ματίας. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μαζί με την τρία τη συμβαστική ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 14. 14. Πέρας ψηφοφορίες. Όχι. Διαμαρτυρία στην αίθουσα. Μισό λεπτό. Δεν πρόλαβα. Λοιπόν, 18-28. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Πέντε συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επτά συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος τις 52 υπέρ κατά αποχές. Κανονικά απορρίπτεται να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά όμως. Παρακαλώ. Πέρασε. 23-26 απορρίπτεται. Τζούρι 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε, Τζούρι. Πώς είπατε? Α, καταπέπτει, καταπίπτει. Άρα λοιπόν, οκτώ συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την εβδομήντα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 24-17 εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζουρι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Καλτέξι 6 υπέρ κατά αποχές, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 6. Κανονικά απορρίπτεται, αλλά για να δούμε. Πέρας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. απορρίπτεται καθαρά. 8.41 δεν σηκώνατε τα χεράκια σας, οπότε δεν είδαμε καθαρά. 76 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάλτε δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάλτ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 24-26 και απορρίπτεται. Τζούρι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτενέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ μισό λεπτό τι είπατε πως είπατε να ελέγξουμε ποιο να ελέγξουμε το 87 87 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ 87 Πέρας. 37-10 εγκρίνεται. Τι είπατε? Να ξαναλέξουμε. Πού είμαστε στην 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές κανονικά απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 90 ηλεκτρονικά. Πέρας. 22-25 απορρίπτεται. 12 υπέρ, ε, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, εντάξει, ελέγχουμε. Το πρώτο μέρος της 149 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 23-26 απορρίπτεται. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 26-24 εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 και 35 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ναι. Τζούρι 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 συμβαστική υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 18 συμβαστική υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Κάλτε 40 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 176 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 19 συμβαστική υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 19. Α, όχι, στην, για 42 ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ναι. 42 ελέγχουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Πέρας. 22-28 και απορρίπτεται. Ζούρι 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζούρι 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177. Τι ελέγχουμε την 176 παρακαλώ. Πέρας. 25-25. Απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 177 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. 19.31. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 180 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Όχι, όχι, συγγνώμη. Την 182 ψηφίζουμε. 182 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα την 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 188. 188 υπέρ, κατά, αποχές κανονικά εγκρίνεται να ελέξουμε όμως ηλεκτρονικά την 188 παρακαλώ. Πέρας. 25-24 εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καλτ 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο. Α, μισό λεπτό. Όχι, 197 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Καλτ 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 215 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 218 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 219, υπέρ κατά χες εγκρίνεται 220, υπέρ κατά χες εγκρίνεται 221, υπέρ κατά από χες εγκρίνεται 222, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 περ κατά αποχές εγκρίνεται 224 περ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέξουμε για την 224 Ποιος ζητάει ηλεκτρονική, ηλεκτρονικό έλεγχο. Ποιος ζητάει. Α, εσείς. 2.24. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 2.24. Πέρας. 10.40. Απορρίπτεται. Καθαρά. 34. Υπέρ. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λυσμονήσαμε τη 2.25. 225 ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζουρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. 44 με 5 αποχές συγχαρτήρια, νομοθετικό ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτελέσματα. 45 υπέρ μία αποχή. Στην αφηματίας συγχαρτήρια. Και τώρα. Πάμε παρακάτω. Σκίνερ, Σκίνερ. Κάτι όμως πρέπει να μας πει ο κύριος, η κυρία Σκίνερ. Κάτι επιθυμείτε παρακαλώ. Σκίνερ, ο κύριος Σκίνερ. Ο κύριος Σκίνερ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σύντομη διόρθωση στον κατάλογο ψηφοφοριών για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει Τροπολογία 28 λέει πως έχει αποσυρθεί. Δεν έχει αποσυρθεί. Είναι λάθος αυτό θα ψηφιστεί και παρακαλώ να το κάνετε αυτό και οι δύο τροπολογίας και 111. Εντάξει και το 28 που δεν απέσαιρε ο εισηγητής. Σκίνερ λοιπόν. Όλα μαζί. Τι. Budget 1, 2, 3 και 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Budget 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 τι γίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 σε δύο μέρες με το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο μέρος. 95-96 και τα δύο μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 98 και 99 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, budget 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 109 Όχι. Από κοινού 107, 108 και 26, αυτές τρεις μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, 110 μαζί με την 27 ήταν. και το 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 Κλοντ. Εμείς είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας. Ψηφίζουμε λοιπόν την 111 αλλά χωρίς ε, προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 113-114 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έχουμε μετά. 115-129 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ 118 είπαμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, μισό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. 118. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 118. πέρα εγκρίνεται. Μπάζε 17 είπ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπάζετ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122. Υπέρ. 122 είπαμε. Ή μήπω παραλείψαμε κάποια. 122, ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ποια έχουμε τώρα την 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες μαζί 39 και 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132, 133, 134 όλες μαζί υπέρ Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να ελέγξουμε κάτι. Τι έχουμε εδώ. Ακούστε, ψηφίζουμε μαζί την 132, την 133 και την 134 και την 136. Ναι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Budget 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Την 137 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 137. 137. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 137. Παρακαλώ. Πέρας. 11.37. Απορρίπτεται. 42. Την έχουν ψηφίσει αυτή. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μαζί τώρα 143, 144, 145 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό. 51, 51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158, 159, 160 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164, 165 μαζί αυτές οι δύο. Α, και η 166 υπέρ. Όχι, όχι, αντιδράσεις. 164 και 165. Αυτές οι δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 τώρα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 166. 166. Πέρας. 22-24 απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πώς είπατε? Όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τροπολογία 4. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 4 παρακαλω Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 39-8. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 budget 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πώς, πώς, πώς, πώς, μισό λεπτό καταπίπτει 81 γι' αυτό πάμε παρακάτω στην 80 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Budget 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές κανονικά εγκρίνεται να ελέγξουμε παρακαλώ 84 ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας 29-18 εγκρίνεται budget 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά α μισό λεπτό αποσύρεται αποσύρεται αποσύρεται αποσύρθηκε 86 13 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 38 υπέρ 5 κατά συγχαρτήρια. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το νομοθετικό ψήφισμα να ψηφίσουμε πρώτα. Ναι, Έχει ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λάθος είναι εδώ. Γιατί λέει, λέει στα αγγλικά στη συνέχεια. Για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις γίνεται λόγος, αλλά εδώ δεν είναι απόφαση. Τι κάνουμε, ψηφίζουμε μόνο το νομοθετικό ψήφισμα, αλλά πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν είμαστε εδώ σε συναπόφαση τελικά, Θα πρέπει να το διορθώσουμε πριν ψηφίσουμε τι λέει η γραμματεία λοιπόν, τι προτείνει. Δύο ψηφοφορίε. Μία για το νομοθετικό ψήφισμα και μία ψηφοφορία τη διαπραγματεύσης. Okay. Ναι, για να δούμε ακριβώ. Ε, νομίζω ότι είναι ακριβέ αυτό που είπατε. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Παρακαλώ. Η ηλεκτρονική ψηφορία, νομοθετικό ψήφισμα. Και αν ψήφισαν όλοι. Εντάξει πέρα 36 36-45. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Και νωρίτερα μάλιστα. Στις 3 ξαναρχίζουμε και πάλι. Σε όλους συγχαρητήρια, καλή ανάπαυση σε όλους και στις 3 και πάλι θα τα ξαναπούμε.